ψηφοφορία για να δούμε αν όλες οι πολιτικές ομάδες δεν υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό. Αρχίζει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Δεν είπα ακόμη ότι έχει λήξει. Ξαναλέω, έχει αρχίσει η δοκιμαστική ψηφοφορία. Τεστ, τεστ, ακόμα είναι τεστ. Γιατί ακόμα δεν έχω πει stop. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τεστ ξαναλέω, ε, δοκιμαστική. Κάποιος δεν είχε ακόμα ψηφίσει. Τώρα κλείνουμε. Εντάξει μου φαίνεται. Προχωρούμε τώρα στην ψηφοφορία. Ψηφίζεται η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διορισμό του κυρίου Βολφ Κλίντς. Όποιος επιθυμεί να Ψηφίσει υπέρ, ψηφίζει ναι. Όποιος επιθυμεί να καταψηφίσει, ψηφίζει όχι. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλες και όλοι. Τέλος, 34 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και 4 αποχές. Άρα, συνιστούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναθέσει τα καθήκοντα στον κύριο Κλίντς και διαβιβάζουμε το σχετικό αποτέλεσμα στην διάσκεψη Προέδρων Πολιτικών Ομάδων. Το επόμενο θέμα της ημερησίας διατάξεως τώρα είναι οι δραστηριότητες και εποπτεία για occupational retirement provisions. Καλύτερα στα αγγλικά παρά στα γερμανικά, λέει ο πρόεδρος, γιατί τα έχω αγγλικά μπροστά μου. Η συγητής μας είναι Brian Hayes. Έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Ξέρω ότι είναι η πρώτη συζήτηση αυτή μετά τη συμφωνία του Συμβουλίου μερικούς μήνες πριν. Επιμέ... Ε, περιμένω να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους σκιώδεις εισηγητές, δεν τους έχω συναντήσει όλους, αλλά περιμένω αυτές τις ε, συζητήσεις και αυτή τη συνεργασία. Τώρα, Υπάρχει και ένα έγγραφο εργασίας ε, για να βοηθήσω τους βουλευτές που μπαίνει σε λεπτομέρειες γύρω από αυτό το θέμα αυτό και ξεκαθαρίζει τα θέματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σωστό να πω ότι υπήρχε μια αρχική άποψη ότι αυτή η πρόταση δεν θα προχωρήσει γιατί θεωρήθηκε αρχικά από την, ε, από την ε, Επιτροπή Γιούνκερ ως έπεσε μάλλον ε, στις περικοπές της, ε, του Better Regulation. Όμως ε, τελικά υπήρξε συμφωνία επί Ιταλικής Προεδρίας το Δεκέμβριο που μας πέρασε και τη συγχαίρω την Ιταλική Προεδρία. Θέλω να σας πω καταρχάς τι γίνεται εδώ. Θέλω να παρουσιάσω το, το πεδίο, το τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τροποποίησε η Κομισιόν αυτή την οδηγία ε, που αρχικά είχε υιοθετηθεί το 2003 και να σας πω και την απόψή μου. Για να... Οι οργανισμοί επαγγελματικών συντάξεων Μισό, λεπτό, Μπράιν, διακόπτω πρόεδρο. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε είναι πολύ δυσάρεστο, ο Φέρμπερ είχε ανοίξει το θέμα αυτό πριν ε, 10 λεπτά. 10 λεπτά πριν από την ώρα που προβλεπόταν. Και ε, θα πρότεινα λοιπόν να κάνουμε μία διακοπή και θα ξεκινήσουμε ακριβώς στις και τέταρτο για να είναι εδώ όλοι οι σκιώδες που τους οποίους δεν βλέπω αυτή τη στιγμή. So, damit machen wir eine Pause bis... Οπότε λέω διακοπή μέχρι τις 4 και τέταρτο. 10 λεπτά διακοπή. Econ Point 9 Reloaded. <laughs> Oder 2.0. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem... Αγαπητοί συνάδελφοι, βλέπω ότι υπάρχουν περισσότεροι τώρα σκιώδεις. Α, για να δω, για να δω. Αλλά εν πάση περιπτώσει έφτασε η ώρα που είχαμε αναγγείλει το θέμα, άρα θα έπρεπε να είναι, είχαν δυνατότητα να είναι. Οπότε, Brian, σε παρακαλώ να επαναλάβεις την εισαγωγή που είχε ήδη ξεκινήσει του θέματο αυτού. Από πλευρά μου να αναφέρω ότι είναι πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Το σχέδιο έκθεσης θα το συζητήσουμε Ιούνιο ή Ιούλιο. Έχουμε λοιπόν χρόνο. Σήμερα είναι η έναξη διαδικασίας. Brian, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ ξανά, Πρόεδρε. Καλό είναι που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για αυτό το σημαντικό θέμα. Καλωσορίζω και τους άλλους κοιόδης συζητητές που ήρθαν εδώ. Μερικές από τις συζητήσεις που είχα μαζί τους ήταν πολύ χρήσιμες, το εκτιμώ. Και θα συζητήσω και με εκείνους που δεν έχω συναντήσει. Είναι μια αρχική συζήτηση όπως σας είπα. Και οι συνάδελφοι θα ξέρουν, Πρόεδρε, ότι μοιράσαμε πριν από δύο εβδομάδες ένα έγγραφο εργασίας το οποίο μπαίνει στις λεπτομέρειες του θέματος. Τα εξηγώ με απλό τρόπο, τι προτείνεται δηλαδή στην, στο κείμενο για τους οργανισμούς επαγγελματικών συντάξεων 2 και αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο συντάχθηκε το κείμενό μου. Ελπίζω οι συνάδελφοι να το βρήκαν χρήσιμο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, είχε προταθεί ότι αυτός ο φάκελος, το IOP 2, δεν θα προχωρήσει η Επιτροπή Juncker στα πλαίσια της καλύτερης νομοθεσίας ε, σκεφτόταν ίσως να μην προωθήσει το θέμα αυτό. Αλλά τελικά η Κομισιόν προώθησε το φάκελο αυτό, δεν τον έκοψε. Και όπως ε, ξέρουν οι συνάδελφοι, το Συμβούλιο ε, συμφώνησε επί Ιταλικής Προεδρίας το Δεκέμβριο για τη γενική προσέγγιση που θα ακολουθήσει αυτό το θέμα. Έχουμε μια πρόταση, έχουμε τη γενική προσέγγιση του Συμβουλίου που είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε τουλάχιστον δύο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τι άποψη έχουν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, θέλω να σα εξηγήσω τι είναι αυτό ο οργανισμό επαγγελματικών συντάξεων, τι είναι αυτό το IORP. Να σα εξηγήσω ποιο είναι το τοπίο των συντάξεων στην Ευρώπη, γιατί είναι μεγάλο θέμα και η συντάξη είναι τεράστιο θέμα. Το IORP είναι ένα τμήμα αυτού του τοπίου. Επίσης θα σας εξηγήσω τι άλλαξε και γιατί η Κομισιόν ε, πρότεινε αυτές τις αλλαγές. Ε, γιατί η πρώτη οδηγία του, των οργανισμών αυτών ήταν το 2003. Να σας κάνω και κάποιες ε, σκέψεις δικές μου για το πού βρισκόμαστε και πώς προτείνουμε να προσεγγίσουμε το θέμα. Ένας τέτοιο οργανισμό είναι ένας οργανισμός επαγγελματικών συντάξεων. Είναι ιδρύματα τα οποία ε, διαχειρίζονται ε, συλλογικά ε, εξ ονόματος των εργοδοτών ε, τις συντάξεις για να δώσουν συντάξεις τους εργαζόμενους. και εντάσσεται στον πυλώνα 2. Ο πυλώνας 1 είναι οι συνεισφορές, οι εισφορές Δηλαδή η σύνταξη γύρατος, ας πούμε, που λέγεται σε ορισμένες χώρες, ε, είναι το βασικό συνταξιδοτικό σύστημα, ας πούμε, που βασίζεται στις ε, εισφορές. Το, έχουμε το πυλώνα 2 που είναι οι επαγγελματικέ συντάξεις και έχουμε και το πυλώνα 3 ε, που είναι οι καταθέσεις, η αποταμίευση που δεν είναι υποχρεωτική από τα άτομα. Έχουμε λοιπόν αυτό το σύστημα σε τρεις πυλώνες και το IORP εντάσσεται στο πυλώνα 2. Υπάρχουν 125.000 τέτοιοι οργανισμοί που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι από αυτούς είναι πάρα πολύ μεγάλοι ε, και αφορούν διάφορες επαγγελματικές ομάδες, ε, μεγάλες εταιρείες. Κάποιοι τέτοιοι οργανισμοί είναι πολύ μικροί, έχουν λιγότερο από 100 μέλη. Επομένως, ε, έχουμε διάφορα, διάφορους οργανισμούς, μεγάλους και μικρούς. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι οργανισμοί και το λέμε αυτό στα έγγραφο εργασία που δημοσιεύσαμε. Είναι ενδιαφέρον που Έχουμε 75 εκατομμύρια Ευρωπαίους που εκπροσωπούνται και 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που διαχειρίζονται αυτοί οι οργανισμοί. Είναι σημαντικό για τον γυράσκοντα πληθυσμό. Και από τον Ιούνιο του 2012 μόνο 84 τέτοιοι οργανισμοί ε, παρέχουν ε, υπηρεσίες διασυνοριακά. Οι περισσότεροι, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία αφορούν μια χώρα. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Ε, να μην πω στους ε, συνάδελφους βέβαια ότι σήμερα στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα λόγω της, ε, των δημογραφικών αλλαγών. Και από το 26% θα περάσουμε στο 53% σε ό,τι αφορά μέσα σε 26 χρόνια στο κατά πόσον εξαρτώμαστε από τη σύνταξη γύρατος. Εάν συνεχιστεί αυτή η τάση, θα έχουμε δύο άτομα που θα δουλεύουν για κάθε συνταξιούχο. Ενώ ήταν τέσσερα. Είναι τέσσερα τώρα. Πώς θα εξασφαλίσουμε αυτές τις συντάξεις. Ε? Αυτό το θέμα θα πρέπει να το δουν τα επιμέρους κράτη-μέλη. Αυτό είναι ευθύνη βεβαίω αρχικά των κρατών μελών ε, σε ό,τι αφορά του τρει πυλώνε 1, 2, 3. Τα κράτη-μέλη έχουν άμεση ευθύνη για να βελτιώσουν τα ταξιδιωτικά συστηματα συστήματα. Κάποια κράτη-μέλη ε, έχουν γενοτομήσει πολύ, ε, κάποια άλλα λιγότερο λόγω των οικονομικών συνθηκών, ε, λόγω τη σύνδεση του πληθυσμού κτλ. Αλλά η οδηγία για του οργανισμού αυτού μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, σημαντικότατο ρόλο, για να υλοποιηθούν να υλοποιηθεί το δυναμικό ε, των οργανισμών επαγγελματικών συντάξεων και να έχουμε και κέρδη λόγω της αποτελεσματικής λειτουργίας αυτών των οργανισμών. Γι' αυτό λοιπόν η οδηγία τροποποίησε την ε, στην οδηγία του 2003. Το 2003 είχαμε την αρχική οδηγία που σας είπα και τότε εστιαζόμασταν στο να μπορούμε οι οργανισμοί επαγγελματικών συντάξεων να υποφελούνται από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων και της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών. Ο βασικός στόχος της οδηγίας ήταν να επιτρέψει μεγαλύτερη διασυνοριακή δραστηριότητα από τους οργανισμούς αυτούς. Τα κράτη-μέλη εφάρμοσαν αυτή τη διάταξη με διαφορετικούς τρόπους όμως και οι περισσότεροι οργανισμοί δουλεύουν σε εθνικό επίπεδο, το είπα αυτό Έχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό ε, διασυνοριακών οργανισμών επαγγελματικών συντάξεων. Ε, η Κομισιόν βλέπει διάφορου λόγου για του οποίου η οδηγία θα πρέπει να τροποποιηθεί. Νομίζω ότι είναι καλό, έτσι για πρακτικού λόγου. Εγώ ήμουνα επί 18 χρόνια στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο και ασχολούμουν με νομοθετήματα. Ε, γενικά, είναι καλή κοινοβουλευτική πρακτική είναι να θεωρούμε την ισχύουσα νομοθεσία και να την επικαιροποιούμε, να είναι κατάλληλη για τους σκοπούς του σημερινού, ας πούμε. Στην πρόταση της Κομισιόν καταρχάς ε, υπάρχουν προληπτικοί φραγμοί για τη διασυνοριακή δραστηριότητα των οργανισμών αυτών αναγνωρίζουν στην Κομισιόν ότι υπήρχε μεγάλη αλλαγή. Ε, από εκεί που είχαμε ε, συντάξεις που να βασίζονται σε ανταποδοτικές συντάξεις σε συντάξεις που βασίζονται σε εισφορές. Η Κομισιόν λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν τα μέλη, ε, πληροφορίες, τα μέλη αυτών των οργανισμών, ε, πληροφορίες ε, λεπτομερείς. Αν ας πούμε, αποφασίσεις να αγοράσεις ένα σπίτι, ε, θα πρέπει να ξέρεις ε, που βρίσκεται αυτό το σπίτι. Ε, είναι σημαντικό να ξέρεις, εν πάση περιπτώσει, αν αποφασίσεις να εργαστείς, ε, αν θα υπάρχει σύνταξη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος, πρέπει, είναι βασικές πληροφορίες, πρέπει να υπάρχουν για τη διαχείριση και τη διαφάνεια που είναι απαιτήσει για τους οργανισμούς αυτούς. Η Συμφωνία του Συμβουλίου έκανε σημαντικές αλλαγές στην αρχική πρόταση της Κομισιόν γύρω από το θέμα των ε, ανταποδοτικών συντάξεων, των ε, ε, διασυνοριακών μεταφορών των δικαιωμάτων και των κατευθυνότητας πράξεων. Ήταν αρκετά επίμαχο θέμα, ειδικά για κάποιο μικρό αριθμό κρατών μελών. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο έκανε, έφτασε σε αυτή τη γενική προσέγγιση και έφτασε στη Συμφωνία Επιταλικής Προεδρίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εκτιμήσουμε. Είναι σημαντικό. Είναι τόσο βέβαια ευαίσθητο το θέμα ε, για κάποια κράτη-μέλη που υπήρχε κόλλημα στην αρχή, αλλά τελικά υπάρχει γενική προσέγγιση. Λοιπόν, τι θέση μπορούμε να πάρουμε. Αναγνωρίζω ότι είναι θέμα καταρχάς των κρατών μελών. Αυτά αποφασίζουν για το συνταξιδοτικό του σύστημα. Θα ήταν λάθος κατά την άποψή μου να έχουμε μία λύση για αυτούς τους οργανισμούς και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε έτσι. Θα πρέπει να καταλάβουμε και να αναγνωρίσουμε ότι οι συστάσεις, η συνταξιδοτική κάλυψη στην Ευρώπη ε, εξαρτάται σε, μεγάλο βαθμό από την αντίληψη που έχει το κάθε κράτο μέλος. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε επίση ότι ιστορικά σε κάποια κράτη-μέλη οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι θεωρούσαν ότι είναι κοινωνική υποχρέωση, ή μάλλον οι εργοδότες θεωρούσαν ότι είναι κοινωνική υποχρέωσή τους να δώσουν σύνταξη στους εργαζόμενου και να είναι καλή η σύνταξή του. Είναι αυτή η ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Γι' αυτό έχουμε αυτές τις, αυτά τα συστήματα συντάξεων. Και οι, τα συνδικάτα έχουν στεναρή άποψη. Δεν θεωρούν ότι είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα απλό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουν ε, όταν πάνω σύνταξη άνθρωποι τα απαραίτητα λεφτά, την απαραίτητη σύνταξη. Ε, επίσης, ε, έχουν μεγάλη επίπτωση αυτοί οι οργανισμοί σε μικρές ε, σε μικρό αριθμό χωρών. Υπάρχουν χώρε που έχουν λίγου τέτοιου οργανισμού. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια επίπτωση. Ε, μην ξεχνάμε την κινητικότητα του, των εργαζομένων στην Ευρώπη. Το 3,5% των εργαζομένων ε, είναι περίπου 8 εκατομμύρια Ευρωπαίοι που κινούνται διασυνοριακά. Ε, και λογικό είναι, λόγω των δημογραφικών αλλαγών που θα υπάρξουν τα επόμενα χρόνια, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι θα αναγκαστούν να πάνε σε άλλο κρατό ε, μέλο για να βρουν δουλειά. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να έχουν επαρκή συνταξιδοτική κάλυψη καθώς θα μετακινούνται ε, από κράτος σε κράτος. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε λοιπόν ότι ναι, είναι μικρός ο αριθμός των χωρών που έχουν τέτοιους οργανισμούς, αλλά για λόγους ανταγωνιστικότητας, για λόγω, κινητικότητας, η ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό εργατικό δυναμικό στο μέλλον θα λειτουργεί διαφορετικά. Και γι' αυτό θα πρέπει ε, να υπάρχουν οργανισμοί που λειτουργούν σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. Είναι λογικό αυτό αν θέλουμε να ενθαρρύνουμε ε, τον κόσμο να μετακινηθεί σε μια άλλη χώρα για να βρει δουλειά. Τρίτον, ένας από τους βασικούς στόχου κατά την άποψή μου, θα πρέπει να είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εσωτερική αγορά ε, των οργανισμών. Έχουμε κάποια κράτη-μέλη που ιστορικά έχουν δημιουργήσει τέτοιου οργανισμού. Ε, δεν θέλουμε όμω να έχουμε πάρα πολλέ ρυθμίσει, κανονισμού κτλ και επίσης να μην αντιγράψει η Κομισιόν τους κανόνες για τις ασφαλίσεις ή για την αφαιρεγγιότητα για τους οργανισμούς αυτούς. Θα ήταν κρίμα. Μετά από την κρίση, πολλοί εργαζόμενοι ψάχνουν να βρουν συστήματα τα οποία είναι ε, φερέγγια ε, και που θα τους δώσουν ε, κατάλληλη σύνταξη όταν συνταξιδοτηθούν το να εφαρμόσουμε τους κανόνες περιφερειακότητας που ισχύουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες θα ήταν λάθος. Και νομίζω ότι η Κομισιόν, η Κομισιόν ε, συμφώνησε ότι θα ακολουθήσει αυτή την οδό. Επίσης, η επικοινωνία είναι σημαντική. Οι εργαζόμενοι είναι σημαντικό να ξέρουν ποια είναι τα συστήματα που υπάρχουν, έχουν δικαίωμα να ξέρουν τι απόδοση θα έχουν, ε, τι σύνταξη θα πάρουν, θα τους δώσουν στο μέλλον και να ε, απαντηθούν σωστά οι ερωτήσεις. Ε, είδαμε σε μερικές ε, χώρες όπως στην Ολλανδία παραδείγματα μοντέλων. Δηλαδή δίνουν πληροφορίες στον κόσμο φτιάχνοντα μοντέλα. Ε, εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν αυτές τι πληροφορίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μοντέλα ως παραδείγματα ε, και σε άλλες χώρες. Χωρί να τα επιβάλλουμε όμως αυτά σε άλλες χώρες. Δεν πρέπει να τους επιβάλλουμε αυτά αυτό το μοντέλο πληροφοριών κατά ανάγκη, αλλά να του το υποδείξουμε. Αυτή είναι η προσέγγισή μου. Και αν το δεχτεί η Επιτροπή μα και οι συντονιστέ, θα πρέπει να κάνουμε μια δημόσια ακρόαση. Νομίζω ότι μπορούμε να την κάνουμε κάποια στιγμή το Μάιο. Εγώ είμαι ανοιχτό σε αυτό το θέμα. Θέλω να ακούσω και τι απόψει των σκιωδών και των υπολείπων ευρωβουλευτών για το πώς θα βελτιώσουμε το κείμενο. Η προσέγγιση μου γενικά όμως είναι να το δούμε με προσοχή, γιατί η συνταξιωτική κάλυψη είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ένας μικρός αριθμός χωρών έχουν ήδη δημιουργήσει ε, ένα πολύ στεναρό σύστημα συνταξιωτικής κάλυψης που πρέπει να το σεβαστούμε. Αυτά για τη γενική συνταξιωτική αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Αυτά και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστώ για την εκτενή εισαγωγή αντί του Πολ Τάγκ η Ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και ο πρόεδρος, θα μιλήσω ε, για λογαριασμό του Πολ, ο οποίος είναι από σήμερα. Εγώ βέβαια το έχω συζητήσει διαμακρών το θέμα μαζί του και θα επαναλάβω μάλιστα και επιλέξει μερικά πράγματα από αυτά που μου ζήτησε να πω. Ο Πολ λέει πρώτον ότι επιθυμεί να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας που, που συνοψίζει τα σημαντικά θέματα για τη συζήτηση. Συμφωνώ με τον κύριο Χέις για να υπάρξουν ε, βιώσιμα IOP στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υποστηρίζει επίσης την παρατήρηση ότι η ευαισθησία του θέματος έχει σχέση με το γεγονός ότι μικρός αριθμός χωρών μελών έχουν δευτερεύοντα συστήματα, συνταξιωτικά συστήματα. επίσης, λέει επίσης ότι η έκθεση σωστά λέει ότι τα ΕΟΠ είναι τα πρώτοι θεσμοί που ε, θα φροντίσουν για τους συνταξιούχους και κυρίως για την απόδοση επενδύσεων για τους ε, δικαιούχους των συντάξεων είτε σημερινούς είτε μελλοντικούς. Επίσης ο συνάδελφός μου ζήτησε να τονίσω ορισμένες ανησυχίες που έχει σχετικά. Το έγγραφο εργασίας του κ. Hayes λέει αναφέρει το γεγονός ότι το Συμβούλιο Μελετών Αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλύσει το θέμα δύο φορές και δεν μπόρεσε να εκδώσει θετική ε, γνωμοδότηση. Ο Πολ θεωρεί ότι αυτό είναι ατυχές και δυστυχώς συμφωνεί με την παρατήρηση του εισηγητού ότι οι ενστάσεις του Συμβουλίου ε, Μελέτης Αντικτύπου εξακολουθούν να ισχύουν. Εκτός από αυτό, το ευρωπαϊκό, το μάλλον ε, η υπηρεσία ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ταχθεί πολύ ε, κριτικά απέναντι στον φάκελο αυτό. Υπάρχει και απουσία μελέτης αντικτύπου και ε, θέτει υπό αμφισβήτηση την ευρωπαϊκή διάσταση των προτινόμενων δράσεων. Ίσως να έχει περάσει ο χρόνος όταν δηλαδή αποκλείστηκαν τα κεφάλαια από την πρόταση ΑΟΙΟΠ, αλλά εφόσον σημαίνει αυτό η Κομισιόν θα έπρεπε να μας είχε ενημερώσει για ποιο λόγο Άραγε απαιτείται η πρόταση. Και εκτός από αυτό ο Σάνφον Πολ λέει ότι δεν είναι σαφές γιατί απαιτείται ανάληψη δράσης τώρα. Η πρόταση δεν περιλαμβάνει καμιά πληροφορία για το προτινόμενο χρονικό πλαίσιο ούτε για τις διάφορες δράσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Και ρωτά αν ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν μπορεί να ενημερώσει περισσότερο στο τέλο δηλαδή τη ανταλλαγή απόψεων των βουλευτών. Ο κ. Στάνγκ λέει επίση ότι ω σκιώδη συζητητή εξακολουθεί να συζητεί το θέμα αυτό με την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ιδίως δε στα πλαίσια της προσπάθειας βελτίωσης της νομοθεσίας, που στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Χέρης προηγουμένως, ο Πολ θεωρεί ότι η πρόταση αυτή δεν ε, ανταποκρίνεται στα ε, υψηλά στάνταρτ που απαιτούνται και δεν δικαιολογείται απαραίτητα η, η, πρότασή της. Ashley Φοξ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή για το πλήρες και χρήσιμο κείμενο που σε μόνο 8 σελίδες μπορεί και συνοψίζει όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουμε. Και αν κάποιος επιθυμεί να μάθει καλά θα κάνει να το διαβάσει. Είναι μια καλή αφετηρία. Και συμφωνώ με τις απόψεις που άκουσα μόλις να μεταφέρονται από τον σκιώδη εισηγητή των σοσιαλιστών για την μελέτη αντικτύπου. Το έχουμε δει δύο φορές το θέμα αυτό, το Συμβούλιο μάλλον μελέτη αντικτύπου και παρόλα αυτά δεν μπορεί να, δώσει, να εκδώσει θετική γνωμοδότηση. Εξακολουθώ να θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητη νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια και την πρόταση δεν την έχει αποσύρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρώ ότι είναι σωστή η προσέγγιση του εισηγητού. Θα υπάρξει συνένεση στην Επιτροπή Οικονομικών να μην προχωρήσουμε. Θα, τότε θα, θα είμαι διατεθειμένο να το συζητήσω. Θεωρώ ότι στόχο τη νομοθεσία πρέπει να είναι η προσπάθεια διευκόλυνση τη λειτουργία τη ενιαία αγορά και η μεγαλύτερη διαφάνεια. Συμφωνώ με τον ότι πρέπει να αποφύγουμε αυτό το ενιαίο μέγεθος για όλους. Τέσσερις χώρες μέλη έχουν διατάξεις IOP που έχουν ένα κοινωνικό σκοπό που ανταποκρίνεται στις διαφορετικές παραδόσεις προστασίας ε, του κόσμου της εργασίας και προσφέρουν ε, ευκαμψία στις χώρες μέλη και ο ΕΟΠ e υποχρεούται να, να δαπανίσει σημαντικούς πόρους χωρίς να υπάρχει ωστόσο σημαντικό όφελος για τις χώρες μέλη. Όσο περισσότερη νομοθεσία φορτώνουμε σε αυτά τα μικρά συνταξιοδοτικά προγράμματα θα καταλήξουμε άνθρωποι που δεν έχουν υψηλά εισοδήματα και δεν μπορούν να έχουν υψηλέ συντάξει, θα έχουν ακόμα χαμηλότερε συντάξει επειδή καλούνται να πληρώνουν το κόστο αυτό. Οποιεδήποτε νέε απαιτήσει λοιπόν θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα υφιστάμενα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Κύριε Πρόεδρε, έχω πέντε ανησυχίες και θα σας τις πω σύντομα. Η απέτηση να όλα τα μέλη δημόσιων υπηρεσιών να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Αυτό σημαίνει να... Αυτό ίσως έχει αφαιρεθεί. Αν αυτό είναι αλήθεια, τότε έχει καλώς. Αλλιώς θα θέλω να σταματήσει, θα ήθελα να σταματήσει. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για υπερβολικές απαιτήσει διαφάνειας, ιδίω για τις δηλώσεις, για τις συντάξεις, που αυτό μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα και μπορεί να σημάνει ε, σημαντική αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μου αρέσει επίσης η αξιολόγηση κινδύνου του τύπου one size fits all. Αυτό πρέπει να δώσει ευκαμψία στις χώρες μέλη για να προσαρμόζουν τις ε, προβλέψεις. Και συμφωνώ επίσης με την προσέγγιση του εισηγητού οποιουσδήποτε τροπολογίες να ακολουθήσουν τη τακτική διαδικασία οι κατεξουσιώτηση πράξεις αλλάζουν το καθεστώς αυτό και θέλω να αφαιρεθεί η σχετική μνήμα. Η συνολική προσέγγιση του Συμβουλίου έχει κάνει πρόοδο εγκρίνοντα την αρχική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει τώρα να βασιστεί στην εργασία αυτή του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου, για να επιτύχει την ιδανική δυνατόν έκβαση για τα ΙΟΠ και τι χώρε μέλη. Ευχαριστώ κύριε Άσλι Άλντε Σοφίντ Φέλντ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα, αλλά προσπαθούσα να πάω σε δύο επιτροπές σχεδόν ταυτόχρονα. Δύο γενικές αρχές που θα πρέπει να μας οδηγούν στη συζήτηση είναι η εξή Πρώτη, όπως είπε και ο εισηγητής, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί βεβαίως. Αλλά παράλληλα δεν πρέπει να έχουμε ταμπού, τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Η όλη ιδέα ότι όλα πάνε πολύ καλά, ιδίως στις τέσσερις χώρες όπου έχει προχωρήσει πολύ το θέμα αυτό, είναι βεβαιασμένη, ε, βεβαιασμένο συμπέρασμα. Και επιπλέον δεν πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση σαν να αφορά μόνο τις τέσσερις χώρες το θέμα αυτό. Είναι ευρωπαϊκή αυτή η πρωτοβουλία. και συμμερίζομαι μερικές από τις προτάσεις της αρχικής οδηγίας και της αναθεώρησης. Για παράδειγμα, να υπάρξει ενιαία αγορά και να καταργηθούν οι φραγμοί και να υπάρχει καλύτερη διαμεθοριακή παροχή τέτοιων υπηρεσιών και να βελτιωθεί και η ασφάλεια της παροχής τέτοιων συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, συντάξεων δηλαδή. Αυτοί οι οργανισμοί Ορισμένοι λένε ότι επειδή έχουν κοινωνικό στόχο δεν θα έπρεπε να συζητιώνται. Μα γι' αυτό πρέπει να το συζητήσουμε, επειδή εξυπηρετούν κοινωνικό στόχο. Στην ε, Ολλανδία έχουμε τέτοια συστήματα οργανισμών παροχή επαγγελματικών συντάξεων, IORP, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτοί οι οργανισμοί δεν έχουν καθόλου προβλήματα. Και αυτό μα το έδειξε η χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχουν κάποια μειονεκτήματα στο σύστημά μα Ναι, μεν θεωρώ ότι είναι θαυμάσιο, αλλά δεν είναι άτρωτο, έχει κάποιες αδυναμίες. Όπως απέδειξε ακριβώς η χρηματοπιστωτική κρίση, τους κινδύνους τους φέρουν δυσανάλογα όλο και περισσότερο οι επόμενες γενναίες. Όταν λοιπόν συζητάμε το σύστημα αυτό, πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε τα ωφέλη να τα συμμεριστούν όλες οι γενιές και έχω πλήρη συνέστηση ότι δυσανάλογα μεταφέρεται το βάρος και η κίνδυνη στις επόμενες γενιές. Και ανησυχώ για την ε, στεναρότητα του συστήματος. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν χρησιμοποιώντας άλλους όρους. Βεβαίως πρέπει να το συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μόνο τα διαμάντια είναι παντοτινά, όλα τα άλλα αλλάζουν. Αλλάζουν και τα συνταξιδοτικά ταμεία και πρέπει να αλλάζουν. Γιατί αλλάζει ο τρόπος εργασίας μας. Δεν αρχίζουν όλοι να δουλεύουν στα 15 πλέον και δεν δουλεύουν για τον ίδιο εργοδότη 40-50 χρόνια. Μπορεί να δουλέψουν για διάφορους εργοδότες, μπορεί να αλλάξουν χώρα, τουλάχιστον θέλουμε να το αυτό, μπορεί να δουλέψουν ως αυτοαπασχολούμενοι για μια περίοδο, μπορεί να σταματήσουν να δουλεύουν για ένα διάστημα. Αλλάζει και γενικά η διάρθρωση της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα της ευρωπαϊκής. Άρα είναι πιστεύω αναγκαίο να τα συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και λυπηρό που στη χώρα μου ορισμένοι αμέσως και φωνάζουν όχι να μην τα συζητήσουμε, όχι να η να μην μπλέκεται η Ευρώπη, να μην μπλέκονται οι Βρυξέλλες, να μην βάλουν χέρι στις συντάξει μας. Μα δεν πρόκειται περί αυτού. Αντίθετα. Εγώ ανησυχώ πολύ περισσότερο γιατί ότι κάνουν τα ίδια τα ταμεία αυτά. Όπως είπα δυσανάλογα μεταφέρουν τους κινδύνου στι επόμενε γενναίε. Σε αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω, όχι ταμπού στη συζήτηση αυτή, όλα είναι προς συζήτηση. Έχουμε ευθύνη έναντι των επομένων γενεών και όχι μόνο των τωρινών συνταξιούχων. Και τέλος, προς τον ε, Μπολ Τάγκ, ο οποίος είναι απόν, ο Ολλανδός συναδελφός μου, αυτά που είπε όπως τα εκφράσατε εσείς, να ανταποκρίνονται σε έναν βαθμό στο ότι τα Ολλανδικά ταμεία έχουν στη δίκησή τους ε, πολλούς εκπροσώπους των πολιτικών εταίρων που παίζουν μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε τα συνδικάτα δεν είναι πια τόσο αντιπροσπευτικά διότι είναι πολύ χαμηλός ο βαθμός συμμετοχής και η μέση ηλικία των μελών των συνδικάτων είναι 56. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των επομένων γενεών και όχι μόνο αυτών που είναι τώρα ταξιδιωτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σοφία, για την ΚΟΕ. Ο Μιγγέλ Λουομπάν Κρέσπο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιγγέλ Ουρμπάν Κρέσπο. Η πρόταση της Κομισιόν προσπαθεί πρώτα απ' όλα να προωθήσει τέτοιου τύπου οργανισμούς οι οποίοι ανταγωνίζονται τα δημόσια συστήματα συνταξιοδότησης που ε, είναι πολύ πιο ευρείας διάδοσης. Βεβαίως, ορισμένες φορές είναι επιτεύγματα των συνδικάτων, ορισμένες φορές ε, κάνουν κακές πρακτικές, δηλαδή ωφελούν κυρίως ε, τους εργαζόμενους με τις υψηλές αποδοχές της επιχειρήσης, άρα δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και λειτουργούν ως οργανισμοί αυτοκεφαλαιοποίησης. Διότι ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς αγοράζουν μετοχές από την επιχείρηση αυτή και δυσχεραίνουν ε, την επίτευξη σύνταξη για όλους. Θα ήταν αναγκαίο λοιπόν να υπάρξει σαφής ρύθμιση που να συμπεριλαμβάνει σωστές πρακτικές. Δηλαδή να είναι υποχρεωτική η κάλυψη όλων των εργαζομένων, ακόμη και των εξωτερικών συνεργατών. Να υπάρχουν συλλογικέ συμβάσει, να μην επιτρέπεται η αυτοκεφαλαιοποίηση κτλ. Επιπλέον, η πρόταση όπω είναι τώρα θεωρεί ότι πρέπει να ισχύει ως βασική ρύθμιση ε, η ρύθμιση που ισχύει στη χώρα προέλευσης και όχι των χωρών όπου καταλήγει η δραστηριότητα. Αυτό στην ουσία είναι ανταγωνισμός προς τα κάτω. Οι διαχειριστές αυτών των ταμείων θα έχουν την τάση να τα δημιουργούν στις χώρες που έχουν τη λιγότερη ρύθμιση. Τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να μπορέσουν να κινητοποιήσουν κεφάλαιο για τις μεγάλες επενδύσεις, για τις ε, υποδομές όπως το πρόγραμμα Juncker. Δηλαδή θα μεταφέρουμε τον κίνδυνο για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις στην τσέπη των εργαζομένων και αυτές είναι ιδιαίτερα ε, κερδοσκοπικές. Θα ήταν πολύ καλύτερα να απαγορευθεί η επένδυση για επικίνδυνες ή περιβαλλοντικά επικίνδυνες επενδύσεις σε προγράμματα τέτοια ή οι επενδύσεις ε, εάν υπάρχουν ηθικές επιφυλάξει. Και θα πρέπει να δούμε συγκεκριμένα τι σημαίνουν όλα αυτά. Και βεβαίως πρέπει να συμμετέχουν οι ελληνικοί εταίροι, οι οποίοι θα πρέπει να αφοληθούν από αυτά τα ταμεία. Αυτοί θα πρέπει να αποφασίζουν με βάση το περιεχόμενο των επενδύσεων και όχι μόνο σε σχέση με ε, την αναμονή θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ πολύ, Μιγέλ. Τελευταίος από τους Κιώδης, για τους πρασίνους. Ο Έκχαουτ, ο Μπάς Έκχαουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον συγητή για το έγγραφο εργασίας για να ξεκινήσει τη συζήτηση. Άκουσα τον πρώτο γύρο σκιωδών και πολλά υπόσχεται αυτή η συζήτηση για να δούμε τι θέλουμε να επιτύχουμε. Και με εκπλήσει λίγο αυτό που είπε ο Σάνθος Πολταγκ μέσω ημών ότι δεν είναι πεισμένος καθόλου μάλιστα γιατί χρειάζεται αυτή η οδηγία. Πραγματικά με εκπλήσει αυτό. Γιατί έχω εντελώ αντίθετη άποψη. Αλλά γνωρίζω ότι είναι και ενδοολανδικο θέμα. Δεν είναι τυχαίο ότι τρει από του έξι είναι Ολλανδοί. Να μην γίνει συζήτηση, δηλαδή Ολλανδο-Ολλανδικό πάρτι. Ξέρουμε ότι στην Ολλανδία είναι πολύ ευρύτερη η επίπτωση. Έχουν 100 δις ε, επενδύσιμα κεφάλαια οι Ολλανδικοί τέτοιοι οργανισμοί. Άρα δεν μπορούν να επενδύσουν μόνο στην Ολλανδία, πρέπει να επενδύσουν και ευρύτερα, άρα έχει επιπτώσει για την ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία αυτό που κάνουν οι Ολλανδικοί τέτοιοι οργανισμοί. Γι' αυτό το συζητάμε εξάλλου. Είναι σαφές λοιπόν αυτό. Δεύτερον, αλλάζει ο κόσμος. Συμφωνώ με τη Σοφίντ Φέλτ. Αν εξετάσετε αυτά τα ταμεία, δεν καθορίζουμε πλέον ε, τα ωφέλη, αλλά τις συνεισφορές. Αν καθορίζουμε τις συνεισφορές, κατόπιν αυτοί που εξαρτώνται από αυτά έχουν δικαίωμα να ξέρουν περισσότερα για το πού θα πάει και τι ωφέλη θα μπορέσουν να λάβουν από τις ε, συνεισφορές τους. Και ξέρουμε ότι αλλάζει ο τρόπος εργασίας. Δουλεύουμε σε όλη μας τη ζωή, δουλεύουμε στην ίδια θέση εργασίας και αυτό έχει επιπτώσεις ε στη λειτουργία αυτών των οργανισμών. Υπάρχουν λοιπόν ε, βάσιμοι λόγοι για ευρωπαϊκή προσέγγιση, αλλά συμφωνώ με τον εισηγητή ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά κανείς δεν νομίζω ότι πρότεινε μεταξύ των σκιωδών ε, παρακινδυνευμένες προσεγγίσεις και ούτε η Κομισιόν. Και αν δείτε και την προσέγγιση του Συμβουλίου δεν μπορεί να θεωρηθεί καν προσέγγιση. Είναι μη προσέγγιση. Σίγουρα δεν συμφωνούμε. Τώρα, επιμέρους. Η Επιτροπή έκανε αυτή την πρόταση με νομική βάση εσωτερικής αγοράς. Δεν είμαι απόλυτα πεισμένος ότι αυτή η πλευρά ενιαίας αγοράς είναι η πιο σημαντική για τους IORP. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ οι IORP να μπορούν να είναι διεθνείς και μια Ολλανδική εταιρεία να μπορεί να δραστηριοποιείται και στην Γερμανία κτλ. Δεν είναι νομίζω η καλύτερη νομική βάση. Αυτό που είναι κρίσιμο για το θέμα αυτό είναι η ασφάλεια και η διαφάνεια για τους καταναλωτές. Αυτά είναι τα θέματα κλειδιά, τα δύο. Αυτά πρέπει να είναι στο κέντρο της προσοχής μας. Τι εννοώ με ασφάλεια. Ξέρω ότι εξαιρούμε τα συνταξιδοτικά ταμεία από τις προϋποθέσεις φερεγγιότητας. Φερεγγιότητα 2 και τέτοια. Αλλά μπορούμε να περιμένουμε τα ταμεία αυτά. Αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε είναι ότι αυτά που ισχυρίζονται ότι θα χορηγήσουν να μπορεί να ελεγχθεί. Να υπάρχει μια ε, αξιόπιστη αποτίμηση του ότι αυτά που ε, υπόσχονται θα μπορέσουν και να τα υλοποιήσουν. Ότι υπάρχουν λοιπόν επαρκείς προϋποθέσεις για να είναι αξιόπιστοι οι ισχυρισμοί του. Γιατί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διαφορετικά τα σωστικά ταμεία από άλλου οργανισμού που παρέχουν ε, ασφάλιση. Θα πρέπει να υπάρχει ε, αξιόπιστη αποτίμηση. Αν δούμε λοιπόν τις διατάξεις για την ασφάλεια, θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι κατάλληλες. Για τη διαφάνεια. Ναι, πιστεύω ότι χρειάζεται καλύτερη εναρμόνιση της άλλου ενημέρωσης. Της ενημέρωσης ιδίως προς τους δικαιούχους. Και συμφωνώ με τον συγκεκριτή, δεν θα πρέπει να κάνουμε μικροδιαχείριση των οργανισμών, αλλά πρέπει η πληροφόρηση που δίνεις να είναι σαφής. Δεν είναι μικροδιαχείριση να το απαιτείς αυτό. Πρέπει να πετύχουμε σωστή ισορροπία. Να πούμε εντάξει, αυτό είναι πολύ ε, υπερβολική συμμετοχή στη διαχείριση, αλλά αυτό είναι απαραίτητη διαφάνεια δεν είναι παρέμβαση στην καθημερινή διαχείριση όπως λένε πολύ συχνά τα στεγιστοτικά ταμεία θα θέλανε να επιβάλλουμε ώστε να τον λιγότερα σε αυτούς γιατί λένε όλα τα κάνουμε πολύ καλά πολύ καλά τα κάνουμε σας παρακαλούμε κύριοι της Ευρώπης μην παρέμβετε αυτό είναι υπερβολικό και η διαφάνεια των επενδύσεων βεβαίω. θα πρέπει να ξέρουμε σε τι επενδύουν αυτοί οι οργανισμοί και γι' αυτό διαφάνεια πολύ ζωτική σημασία δεν θα σας εκπλήξει ότι εφόσον είμαι πράσινος Φυσικά μας ενδιαφέρει το άρθρο 29. Όταν υπάρχει αποτίμηση του κινδύνου για το μέλλον, να λαμβάνονται υπόψη και οι κίνδυνοι κλιματικής αλλαγής. Κοιτάξτε, ξέρω σας κουράζω, αλλά μιλάμε για σταξιωτικά ταμεία και για τις μελλοντικές γενιές. Εάν τα σταξιωτικά ταμεία επενδύουν σε προγράμματα που έχουν μακροπρόθεσμους κινδύνους θα πρέπει να το ξέρουν οι καταναλωτές. Η διαφάνεια γι' αυτό πρέπει να είναι σημείο κλειδί. Ιδιαίτερα για τα στρεξοδοτικά ταμεία τα οποία κάνουν επενδύσεις ιδιαίτερα μακροπρόθεσμες για τις επόμενες γενιές. Δεν θα πρέπει να αποδώσουν οι επενδύσεις τους για πέντε χρόνια, αλλά για πολλές δεκαετίες. Είναι πολύ ζωτικό. Άρα θα πρέπει να περιμένετε από πλευρά μα ότι θα υποβάλουμε τροπολογίες όπου θα μιλήσουμε για την κατάργηση των επενδύσεων σε ε, οικονομία υψηλής ε, παραγωγής άνθρακα, ε, οξυδίων του άνθρακα. Πρέπει να το συμπεριλάβουμε και αυτό στη συζήτηση. Θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και προσβλέπω στη συνεργασία με την Άσλη. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά σημεία, αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, προσεκτικοί, όλοι συμφωνούμε σε αυτό, αν υπάρχουν σκόπιμοι λόγοι γιατί η Ευρώπη πρέπει να εξετάσει τις επιπτώσεις λειτουργίας των σταξιωτικών ταμείων. Έχει ευρία ενωσιακή επίπτωση λειτουργία τους και οι δικαιούχοι που συμβάλλουν σε αυτά τα ταμεία πρέπει να ξέρουν ότι είναι μακροχρόνια ασφαλή αυτά τα ταμεία και να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία τους. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά και τώρα ποια θα είναι η νομική βάση δεν είναι τόσο σημαντικό. Προσβλέπω στη συνεργασία Σίγουρα θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από αυτού. Να είναι ενωσιακή συζήτηση και όχι μόνο για κάποιες χώρες που έχουν πολλούς τέτοιους οργανισμούς. Σας ευχαριστώ Μπάς. Και να μην είναι μόνο ενδοολανδική συζήτηση. Πάντως έγινε συζήτηση τώρα και εκτός ε, σκιωδών. Τώρα, εκτός των σκιωδών συζητητών, πρώτος ο Τόμας Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως δεν είναι μόνο οι Ολλανδοί που έχουν σχέση με τις συντάξεις, που δίνουν οι επιχειρήσεις, δηλαδή ιδιωτικές συντάξεις, και στη Γερμανία παίζει σημαντικό ρόλο και μιλούμε για 460 δισεκατομμύρια. Ξέρω μερικούς Έλληνες που θα χαίρονταν πολύ αν μπορούσαν να πάρουν κάποια από τα χρήματα αυτά. Συζήτηση που είχε διεξαχθεί τότε αγαπητή Σοφή, μιλείς ε, και δικαίως για το τότε, όμως εδώ τα επιχειρηματικά συμβούλια είναι διαφορετικά. Αυτό που λες πόσο δύσκολο είναι για τους ε, νέους, γιατί χρειάζονται εξασφάλιση για το μέλλον κτλ. Αυτό δεν έχει σχέση με τη σύνταξη γύρατος. Τώρα οι, οι συντάξεις που δίνουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι κάτι διαφορετικό και στη χώρα μου αυτό που γίνεται βασίζεται σε μια συνένεση όπως και για τις κάτω χώρες. Πάντοτε περιλάβαμε στη Γερμανία τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι κοινό έργο αυτών είναι λοιπόν ηθελημένο, είναι επίτηδε. και είναι σημαντική η προσέγγιση αυτή. Προδιετίας είχα συντάξει τη σχετική έκθεση εδώ, σε την εδώ την Επιτροπή ΕΚΟΝ. 44 είχα πει ναι και μία αποχή και, ένας, και μία ψήφος κατά. Άρα ήταν μεγάλη συνεργασία, Ελπίζω να πετύχει το ίδιο ε, αγαπητέ Χέις. Είχε υπάρξει μια διαφορά τότε βέβαια. Εμείς είχαμε προσέξει στο άρθρο 50, δηλαδή είχαμε, είχαμε λάβει δικές μας αρμοδιότητες και αλλού υπήρχαν βεβαίως και σε άλλες ε, υπήρχαν αρμοδιότητες και άλλων επιτροπών, δηλαδή της Επιτροπής Απασχόλησης, στην οποία επίσης συμμετέχω. Τώρα το ότι η Κομισιόν ξανακαταθέτει την πρόταση αυτή, αυτό με παραξενεύει πραγματικά κάπως. Είχαμε πει τότε ότι το σημαντικότερο όλων είναι οι κανόνες φερεγιότητας να μην μπουν μέσα σε αυτό το σύστημα. Ήταν σωστό αυτό. Και θεωρούσα εγώ ότι ο Ζαν Κλοντ Ιούνκερ και άλλοι θα ήταν διατεθειμένοι να πούνε ότι δεν θα το βάλουμε πάλι στην ημερήσια διάταξη. Με την έκθεση σου, Μπράιαν, τονίζεις ποιος είναι ο λόγος για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξαναλέει ότι πρέπει να τεθεί το θέμα στην ημερησία διάταξη. Το Συμβούλιο είχε εκφράσει μεγάλες αμφιβολίες. Μεταξύ άλλων και διότι έχουμε διαφορετικές εμπειρίες. Μην το λησμονούμε αυτό. Έχουμε πολύ ισχυρά συνταξιοδοτικά συστήματα σε κάποιες χώρες και πάρα πολύ ασθενή σε άλλα. Αυτή είναι η διαφορά. Το πλονέκτημα είναι ότι μπορούμε να διδαχθούμε μεν από τους δε. Δεν είναι τόσο η ιδέα της σύνταξης που ε, πλήττονται κιόλας από την πολιτική μηδενικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πώς να επενδύσουν κάποια χρήματα. Εγώ ελπίζω ότι Κάποια χρήματα που μπορούν να επενδυθούν με ασφαλή τρόπο θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν επενδύσεις και μέσα στα πλαίσια του σχεδίου επενδύσεων Juncker. Να πάρουμε δηλαδή τις δυνατότητες για την εξασφάλιση των ιδιωτών επενδυτών, επιχειρήσεις και συνταξιωτικά ταμεία κλπ. να μπορέσουν να επενδύσουν χρήματα εκεί όπου πραγματικά αξίζει. Άρα τα έργα τα οποία θα υποστηριχθούν θα πρέπει να είναι χαρακτήρα βιώσιμου με εξασφαλισμένο μέλλον. Αυτό πρέπει να το εξασφαλίσει και η Κεντρική Τράπεζα. Και ελπίζω να καταλήξουμε σε καλές αποφάσεις. Και ένας παράγοντας, η εξασφάλιση απέναντι στην αφαιρεγκαιότητα. Εμείς και στη μεγάλη κρίση, νομίζω μόνο σε δύο συνταξιωτικά ταμεία υπήρξε η διαδικασία καθάρισης, Όλοι οι άλλοι τα κατάφεραν. Επομένω, η εξασφάλιση κατά τη αφαιρεγκαιότητα είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο Μα έχει επιτρέψει να προχωρήσουμε. Και κάτι ακόμα, το οποίο για μένα εξακολουθεί να είναι ασαφέ. Δεν το κάνουμε για να αλυσοδέσουμε τους εργαζόμενους, να πούμε μείνετε στην επιχείρηση για να εξασφαλίσετε την σύνταξη κτλ. Δεν είναι τόσο σημαντικό αυτό. Θέλουμε για παράδειγμα στη χώρα μου να πετύχουμε κάτι το οποίο τότε είχαμε δει να το αντιμετωπίζει αμήχανα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε πίστη στην επιχείρηση. Δεν θέλουμε job hoppers να φεύγουν από μια επιχείρηση στην άλλη, να παίρνουν δηλαδή τα ωφελήματα από εδώ και από εκεί. Θέλουμε αυτοί οι οποίοι έχουν και τα ποιοτικά προσόντα να μπορούμε να πούμε ότι εξασφαλίζουν και ε, την σταξιωτική κάλυψη. Solvency 2 λοιπόν, όχι, να μην μπει μέσα. Ελπίζω να παραμείνει αυτό. Συμφωνώ βέβαια με τη θέση του Ashley Fox για την εκτίμηση των επιπτώσεων, δηλαδή τη μελέτη που κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Και το σημαντικότερο είναι για τις εξουσιοδότηση πράξη, να αποφασίζει κάποιος δηλαδή για λογαριασμό μας. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε, διότι καταστρατηγούνται έτσι οι δημοκρατικοί θεσμοί. Και τελευταίο, διαφάνεια. Όπως είπαν και οι πράσινοι, Πού γίνονται οι επενδύσεις, πώς, ποια πράγματα επιτυχαίνουν, επιτυχαίνουν οι επενδύσεις. Εγώ έχω κάνει σταδιοδρομία στη διαφήμιση και δεν είχα καν ε, ε, συνταξιοδότηση. Ελπίζω άλλοι να μπορέσουν να τα αποφύγουν αυτό. Αναμένω λοιπόν με ενδιαφέρον τη συζήτηση αυτή που δεν θα διεξαχθεί μονάχα βέβαια ε, μόνο μεταξύ των ε, σκιωδών εισηγητών, αλλά πάντως και διμερώς θα σας δω, έχουμε δώσει ραντεβού, στις ακροάσεις. εφόσον έχουμε και τους διάφορους εταίρους, να φέρουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν σημαντική εμπειρία με τις, συντάξεις, με τις συντάξεις. συντάξει. Βεβαίω, όπως είπε και ο Σοφίνφελτ, μόνο τα διαμάτια είναι παντοτινά. Ε, χρειάζεται ευελιξία και αυτήν πρέπει να δείξουμε. Και αυτό θα επιτρέψει και συλλογή εμπειρίας και από αυτούς οι οποίοι δεν έχουν ακόμα σχετική εμπειρία με τέτοια συστήματα. Ευχαριστώ κύριε Μάνη. Φέλτ ζητεί πάλι το λόγο. Ευχαριστώ. Να μην υπάρχει μια παρεξήγηση, ε, αγαπητέ Τόμας. Είπες ότι οι οργανισμοί δεν έχουν καμία σχέση με την ε, διάσταση που αφορά τις διάφορε γενιέ. Όμω έχουν. Οι νέοι πληρώνουν σε ένα συνταξιδοτικό ταμείο που με τη σειρά του δίνει συντάξει ε, στα μέλη του, στου δικαιούχου. Και είναι και υποχρεωτικό αυτό το σύστημα. Προφανώς πρέπει να μιλάμε για το θέμα των γενναίων εδώ. Δεν μπορούμε να σκεφ... ισχυριστούμε ότι αφορά μόνο τον πρώτο Όχι, αφορά και τα συστήματα του δεύτερου πυλώνα. Εσύ λες ότι δεν σ' αρέσει το να αλλάζουμε επιχείρηση, από, να πηγαίνουμε από επιχείρηση σε επιχείρηση. Όλα αυτά τα θέματα καθορίζουν την καριέρα ε, των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα πρέπει να επιλέγουν ίδια την καριέρα τους, αλλά ό,τι και να αποφασίσουν, είτε τους αρέσει να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο επιχείρηση ή, ή αποφασίσουν να δουλέψουν σε όλη την καριέρα στον ίδιο εργοδότη. Το θέμα είναι να πάρουν ε, σωστή σύνταξη, καλή σύνταξη στο τέλο. Και όλοι, είτε είναι 21 ε, χρονών, είτε 71, όταν ε, φτάσουν τη σύνταξη, το θέμα είναι να πάρουν σωστή σύνταξη με βάση τις εισφορές τους. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό οι νέοι, αυτό είπα εγώ, να πλέον δυσανάλογα στο ταμείο και αυτά που θα πάρουν όταν φτάσουν σε ηλικία συνταξιοδότηση να μην είναι τόσα όσα είναι σήμερα ηλικιωμένοι, όσα παίρνουν οι σημερινοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι αποφελούνται πολύ περισσότερο και παίρνουν υψηλότερε συντάξει από αυτέ που θα πάρουν οι μελλοντικοί ηλικιωμένοι. Να το, να συζητήσουμε λοιπόν αυτό. Δεν βλέπω κανένα άλλο να θέλει το λόγο. Α, η Αναλή Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ανησύχησα κάτι διάρκεια τη συζήτηση λιγάκι. Προφανώ εγώ προσωπικά ε, συμμερίζομαι πολλές από τις ανησυχίες του Πολ. Όχι γιατί θέλω να υπερασπιστώ συγκεκριμένα συμφέροντα ή τους μεγάλους εργοδότες ή τα συνδικάτα κτλ. Όχι καθόλου για αυτό το λόγο. Παρότι με χαρά σας λέω ότι εγώ είμαι μέλος ε, συνδικα... ενός συνδικάτου όπως και εκατομμύρια άλλων εργαζομένων της χώρας μου. Αλλά Αυτά τα, αυτοί οι οργανισμοί επαγγελματικών συντάξεων ε, τα έχουν πάει πολύ καλύτερα σε ορισμένε από τις χώρες μας και γι' αυτό ε, και ειδικά όταν είναι ιδιωτικοί και πρέπει να αναγνωρίσουμε αυτό. Εγώ ως μέλος ενός μεγάλου οργανισμού το αναγνωρίζω. Χρησιμοποίησε τους μηχανισμούς, τους κυβερνητικούς, τους κρατικούς δηλαδή, για να εξασφαλίσει μια σωστή διοντολογική ε, επενδυτική πολιτική. Ε, αυτό το κάνει το, ένας κρατικός οργανισμός αντίθετα με αυτό που κάνουν ε, κάποιοι ιδιωτικοί οργανισμοί. Και συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που είπατε για το θέμα των, των συστημάτων. Πρέπει πρέπει να συζητήσουμε θέματα που δεν έχουμε αγγίξει σήμερα. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ε, ανάμεσα στα δύο φύλλα στι συντάξει. Διαφορετικέ συντάξει παίρνουν οι γυναίκε και διαφορετικέ άντρε. Να μην πάμε το. να μην μετακινήσουμε το βάρο που δίνουμε σε αυτού του οργανισμού, κρατικού οργανισμού επαγγελματικών συντάξεων και να δώσουμε το βάρο στου ιδιωτικού οργανισμού. Όχι. Μην ξεχνάτε ότι αυτό είναι τμήμα του κοινωνικού ιστού σε διάφορα κράτη-μέλη. Επομένως θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα προχωρήσουμε και να αναγνωρίσουμε τι, ποιο σύστημα έχει καλές επιδόσεις και ποιο σύστημα έχει κακές επιδόσεις. επιδόσεις. Ε, και επιπλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλοι οι stakeholders να εμπλακούν. Ε, στο παρελθόν ο Πόλη είχε εμπλακεί σε αυτές τις συζητήσεις ε, και πιστεύω ότι πρέπει να ξαναρχίσουν αυτέ οι συζητήσει. Γιατί αυτοί οι κοινωνικοί εταίροι, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε παλιέ συζητήσει, έχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούν και μην ξεχνάμε ότι εκπροσωπούν εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ, Ανελίζε. Να κοιτάξω το ρολόι. Έχουμε 10 λεπτά ακόμη που μας για να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάλι τον εισηγητή αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο επ' αυτού. Ο κύριος Βίσνερ λοιπόν από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ για το κείμενο που υπέβαλε ο εισηγητής. Δεν έχουμε σχόλια. Νομίζω ότι είναι μια σωστή ανάλυση της κατάστασης. Πολλά σχόλια έγιναν. Πολλά μας βρίσκουν σύμφωνους. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει νέα οδηγία IORP 2. Υπάρχει η οδηγία IORP 1 υπήρχε διότι θέλαμε να υπάρχει διασυνοριακή δυνατότητα λειτουργίας και μία ελάχιστη προϋπόθεση διακυβέρνησης και διαφάνειας. Πρέπει να θέσουμε λοιπόν το ερώτημα. Αρκεί αυτή η οδηγία, μήπως μπορεί να βελτιωθεί. Και βεβαίως έχουν υπάρξει και εξελίξεις που μας όθησαν στο συμπέρασμα ότι είναι κατάλληλη στιγμή για να βελτιώσουμε την κατάσταση πρώτη εξέλιξη αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας και κάποια ταμεία ήθελαν να μπορούν να λειτουργήσουν διεθνώς. Άρα υπάρχει μια τάση για πιο διεθνή λειτουργία. Επίσης μια τάση που διαπιστώσαμε είναι ότι σε κάποια κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι οργανισμοί ήθελαν να μπορούν να τα εισαγάγουν. Ήθελαν λοιπόν ε, βοήθεια και ήθελαν να ξέρουν εάν θα είχε να δημιουργήσουν τέτοιους οργανισμούς ή να αντιγράψουν οργανισμούς που λειτουργούν καλά σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτός είναι ένας από τους κυρίους λόγους γιατί υπήρξε συνενετική άψη του Συμβουλίου τελικά. Γιατί η συζήτηση δεν αφορούσε μόνο τις 4-5 χώρες που ήδη έχουν IORPs, αλλά υπήρχε πολύ ενδιαφέρον από άλλες χώρες που δεν έχουν τέτοιους οργανισμούς και θα ήθελαν να δημιουργήσουν. Είναι λοιπόν ευρωπαϊκή συζήτηση. Πολύ σημαντικό να την αντιμετωπίσουμε έτσι και να έχουμε τέτοιους οργανισμούς σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη-μέλη που να λειτουργούν σωστά. Αυτή λοιπόν η οδηγία IORP2 μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Τώρα επιμέρους για πιο επικριτικές παρατηρήσεις που ακούσαμε για την κοινωνική διάσταση. Η πρόταση της Επιτροπής θέτει το θέμα της λειτουργίας και των κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τη λειτουργία. Δεν αμφισβητούμε τον τρόπο λειτουργίας. Η διακυβέρνηση είναι θέμα γιατί κάποιοι εμπειρογνώμονε σε αυτού του οργανισμού μπορούν να κάνουν τη δική του αποτίμηση κινδύνων. Βεβαίω αυτό έχει μια κοινωνική διάσταση. Αλλά αν θέλετε να υπάρχουν κοινωνικέ επιπτώσει, πρέπει να επιτύχουν την απαραίτητη απόδοση αυτοί οι οργανισμοί. Άρα πρέπει να υπάρχει μια προληπτική οικονομική διαχείριση. Δεν έχει καμιά πρόθεση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αμφισβητείτε τον τρόπο λειτουργία των οργανισμών που έχουν αυτή την κοινωνική διάσταση. Θέλει να διασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή ρύθμιση στη λειτουργία του. Αυτό το Συμβούλιο Αποτίμησης Κινδύνων. Αποτίμηση επιπτώσεων. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την πρόταση. Αυτή είναι η πρώτη μου απάντηση. Ως Επιτροπή. Ο δεύτερος λόγος που προτείνουμε αυτό το Συμβούλιο είναι γιατί θέλουμε να έχουμε στοιχεία για το πώς θα αλλάξει η κατάσταση στο μέλλον. Ξέρουμε ότι κάποια τέτοια ταμεία θέλουν να έχουν διεθνή συνεργασία Δεν ξέρουμε όμως πόσους τέτοιους οργανισμούς θα έχουμε σε 10 χρόνια. 50, 10.000. Ξέρουμε λοιπόν πως είναι αδύνατο να έχουμε στοιχεία τώρα για το μέλλον. Αλλά χρειάστηκε να πάρουμε μια απόφαση. Έχει μια πολιτική διάσταση όπως το Συμβούλιο. Σε τελευταία ανάλυση είναι μια πολιτική απόφαση με βάση τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε, ό,τι είναι διαθέσιμο. Σας καλούμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την πολιτική ζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Δίσνερ. Ε, πάλι ο Μπράιν Χέις ο συζήτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους καθώς και σκιώδεις συζητές για την συζήτηση πολύ καλή αφετηρία συζήτησης στην πρόταση. Και βέβαια ο Τόμας Μαν το 2003 ήταν ο εισηγητής που είχε προωθήσει την πρώτη εκείνη εισήγηση για το ESP1, IORP1. Είχε πετύχει τότε 44 ψήφους υπέρ, μία κατά, δεν ξέρω αν θα πετύχω το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά βεβαίως αναγνωρίζω την επιτυχία του. Πρέπει να πούμε σωστή πράγματα, σκέψεις που μου προκαλούν τα όσα άκουσα. Όταν μιλούμε για συστήματα επαγγελματικών συντάξεων, μιλούμε βέβαια για εργοδότες οι οποίοι συνεισφέρουν στα συστήματα αυτά, αλλά μιλούμε και για τους εργαζόμενους, οι οποίοι και αυτοί αφιερώνουν σε μηνιαία βάση και σε εβδομαδιαία βάση στα ίδια προγράμματα. Δηλαδή πρόκειται για παρετούνται δηλαδή από ένα μέρος των απολαβών τους υπέρ μιας μελλοντική σύνταξη. Άρα υπάρχει μια εταιρική σχέση μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Βεβαίω και χρειάζεται γνωμοδότηση γιατί αυτό περνά μια πολιτική απασχόληση τη αποφάσεις των εργαζόμενων, τι θα κάνουν, πού θα πάνε, αποφάσεις για το μέλλον τους, διότι τα ίδια τους τα χρήματα μπαίνουν στο συνταξιωτικό σύστημα. Άρα για τους απασχολούμενους είναι σημαντικό να έχουν εμπιστοσύνη στο σύστημα στο οποίο συμμετέχουν είτε είναι σε βάση επαγγελματικού κλάδου είτε σε μια επιχείρηση μικρή ή μεγάλη είναι σημαντικό να γνωρίζουν τα πρόσωπα αυτά οι απασχολούμενοι δηλαδή σε τι επενδύουν ως τμήμα του συνταξιδοτικού συστήματος γιατί αναλαμβάνουν μια δέσμευση για το μέλλον για να έχουν κάποιες απολαβές όταν θα φτάσουν σε κάποιο χρονικό σημείο της ηλικίας τους. Είναι λοιπόν κρίσιμο να υπάρχει διαφάνεια σχετικά με το τι συνεισφέρουν και που πάνε τα χρήματα αυτά και συμφωνώ με τους συναδέλφους που έθεσαν το θέμα αυτό και τι ακριβώς κάνουν τα συνταξιωτικά συστήματα. Ανεξαρτήτως αυτού υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες έχουν φτιάξει πολύ ε, περίπλοκα συστήματα επιτήρησης με ombudsman, με ανταλλαγή πολλών πληροφοριών και ούτε καθεξής. Και ορισμένες χώρες που δεν το έχουν πράξει αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δοξάζω τις χώρες εκείνες ή τις χωρίζω σε καλά και κακά παραδείγματα, λέω ότι μπορούμε να μάθουμε εμένα από τους δε και συμφωνώ με τους συναδέλφους που τα είπαν αυτά τα πράγματα, μπορούμε να διδαχθούμε από τις εμπειρίες των άλλων σε ό,τι αφορά το τι έγινε και συμφωνώ με την Σοφή ότι δεν θα πρέπει να, υπά, να, παραμείνει μια υπόθεση 4-5 χωρών που θεωρούν απλά ότι είναι αυτή αποκλειστικά η συνεισφορά τους στο θέμα η συνταξιωτική κάλυψη δεν πρόκειται να εξαφανιστεί ως θέμα είτε του πυλώνος 1, όπου τίθεται βεβαίω τεράστια θέματα λόγω των μεγάλων ελλημάτων, είτε διότι τα κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα των, ε, του πυλώνα 1 δεν αντέχουν, αλλά θα πρέπει να έχουμε τη φιλοδοξία για όλους τους χρήστες ότι μπορούν να αναμένουν να λάβουν κάποτε μια επαγγελματική σύνταξη. Και γι' αυτό συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν θέσει υπόψη μας. Να δούμε δηλαδή, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο να μην είναι γραφειοκρατικό, το οποίο να μην συνεπάγεται πρόσθετο κόστος, συμφωνώ απόλυτα με τον Ashley Fox, ένα σύστημα το οποίο θα ενθαρρύνει όλο και περισσότερα η ΕΣΠ, IORP και διαμεθοριακά και όλα ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει βεβαίως τα τελευταία 12 χρόνια να το πετύχουμε αυτό. Να είναι η μεγαλύτερη φιλοδοξία λοιπόν για όλους τους χρήστες ανεξαρτήτως ε, σε ποια χώρα μέλος ζουν και δραστηριοποιούνται. Τα λέω αυτά διότι δεν θέλω ιδίω στις χώρες εκείνες που έχουν ένα ιστορικό ε, Επαγγελματικών Συντάξεων να αντισμονηθεί το σημαντικό και επιτυχημένο έργο που γίνεται εκεί. Άρα ούτε να υπάρξει ιδέα ότι α, δεν αμφισβητούμε καθόλου, δεν συζητούμε καθόλου τα όσα γίνονται. Ξέρω από τους Ολλανδούς ότι γίνεται ε, μια βαθιά μελέτη και ανάλυση του συστήματός τους ότι έχουν υπάρξει και αρνητικές επιπτώσεις, αρνητικές εμπειρίες με βάση το σύστημα αυτό. Και αυτό πρέπει να κάνουμε. Μιλήσατε και για, την, για τις επενδύσεις και ο Μπάς Εκχαουτ επίσης των πράσινων, εγώ βλέπω ότι εκεί κρύβονται κάποιες ευκαιρίε με στο θέμα, να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή οικονομία με μακροπρόθεσμε μακρόχρονε επενδύσει στα πλαίσια του σχεδίου Juncker, να διαθέτουμε την διαφάνεια και τι πληροφορίε για το τι πράττουν τα συνταξιοδοτικά συστήματα έτσι ώστε και οι άνθρωποι να έχουν κάποια ασφάλεια ότι τα χρήματα που συνεισφέρουν στα συστήματα αυτά θα αποδώσουν ορθά. Βρήκα λοιπόν ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα πρόεδρε. Το λέω προς την κατεύθυνση όλων των συναδέλφων μου, ιδίως βέβαια των σκιωδών εισηγητών. Είμαι ανοιχτό, η προσέγγιση μου είναι ανοιχτή απέναντι στο θέμα αυτό. Θα συνεργαστώ με όλε και όλου του συναδέλφου για το επόμενο βήμα τη πρόταση που είναι να διεξαχθεί δημόσια ακρόαση, εάν συμφωνήσει βέβαια η ε, Επιτροπή Οικονομικών. Να διεξαχθεί λοιπόν μια χρήσιμη συζήτηση και να προχωρήσει έτσι το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μπράιαν. Στην συνέχεια, βλέπω θα ξαναδούμε στις 15-16 Εβδόμου το σχέδιο εκθέσεως προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών τον Σεπτέμβρη και ψηφοφορία, σύμφωνα με το ισχύον χρονοδιάγραμμα, για την ώρα δηλαδή, θα τα ξαναπούμε τον Νοέμβρη. Έχουμε λοιπόν αρκετό χρόνο μπροστά μας για τη διεξαγωγή μιας εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης που είδαμε την αφετηρία της σήμερα. Θα ήθελα να περάσουμε τώρα στο θέμα 4 της ημερήσιας διάταξης το οποίο είχαμε κρατήσει investment, shops and growth και υπενθυμίζω εδώ έκτο, έκτη έκθεση συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εδώ θα συνταχθεί έκθεση. Εμείς δε ως Επιτροπή ΕΚΚΟΝ πρόκειται να εκδώσουμε γνωμοδότηση σήμερα. Θα συζητήσουμε εδώ τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον Κώστα Μαυρίδη των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που είναι εισηγητής. Κώστα. Thank you, Chairman. Should I give a couple of minutes for the people to... Να αφήσω δύο λεπτά για να βγουν... Ε, εντάξει. Υποβλήθηκαν συνολικά 80 τροπολογίες. Δεν θα τη συζητήσω αναλυτικά. Θα εστιάσω σε θέματα, στα θέματα με τα οποία ασχολούνται. Πρώτον, να σχολιάσω μία τροπολογία που υπέβαλε ο κύριος Καρίς, που σωστά υπογραμμίζει ότι ο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβάνει το στόχο της προώθησης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και αλληλεγγύης των κρατών μελών. Και υπάρχει ένας ε, πολύ βάσιμος λόγος γιατί ξεκινάω με αυτό. Διότι αν το λάβουμε αυτό υπόψη, και αυτό δεν έχει αλλάξει δηλαδή, τότε η αλληλεγγύη και η αποτελεσματικότητα πρέπει να είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Πρέπει λοιπόν να καταστεί σαφές ότι ορισμένε τροπολογίε μπαίνουν σε τόσε λεπτομέρειες τεχνικές που υπερβαίνουν το πλαίσιο αυτής της γνωμοδότηση. Δεύτερον, πολλοί προτείνουν ε, διαγραφές. Για παράδειγμα, η τρίτρα επενδύσεων προτείνεται να απαλληφθεί. Προτείνεται να απαλληφθεί η συγχρηματοδότηση των διαφθορτικών και επενδυτικών ταμείων της Ένωσης, ο υπολογισμός των ελλημάτων, για, τη σταθερότητα, για το Ταμείο Σταθερότητας, το Σύμφωνο συγγνώμη, Σταθερότητας και Ανάπτυξης και διάφορα άλλα θέματα. Και παράλληλα υπήρξαν τροπολογίες για το ρόλο των επιχειρήσεων και των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων. Με όλα αυτά υπόψη, ομολογώ ότι περιμένω τη συζήτηση των σκιωδών αύριο αλλά πρέπει επίσης να σας πω πως θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμβασμούς για όλα αυτά τα θέματα γιατί μερικές τροπολογίες είναι πολύ αντιφατικές δηλαδή ε, αντιτιθέμενες για τα ίδια θέματα εκφράζουν πολύ διαφορετικές απόψεις. Επίσης, να διευκρινίσω το εξής. Οποιαδήποτε άποψη ή γνωμοδότηση για την πολιτική συνοχή και την αλληλεγγύη πρέπει να καθιστά απόλυτα σαφές σε οποιοδήποτε τέτοιου τύπου κείμενο ότι η πολιτική συνοχή αφορά όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις ε, περιφέρειες. Αλλά παράλληλα είμαστε εν μέσω κρίσης και πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες περιφέρειες και κάποια κράτη-μέλη έχουν φυγεί περισσότερο από αυτήν την κρίση. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και εφόσον ε, αναφερόμεθα στην πολιτική συνοχή πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις. Τι εννοώ. Όλοι ξέρουμε ότι κάποιες περιφέρειες έχουν πολύ ψηλή ανεργία. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Δεν μπορούμε να γενικολογούμε. Εν πάση Επαναλαμβάνω. Θεωρώ ότι για όλους μας είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε μια ειλικρινή συζήτηση αύριο στη συνάντηση των σκιωδών και ελπίζω να υπάρξει συμφωνία επί πολλών συμβιβασμών ούτως ώστε να εγκριθούν διατυπώσεις για πολλά θέματα που όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτή τη γνωμοδότηση. Όμως, παράλληλα πρέπει να τονίσω το εξή. Για ορισμένα σημεία θεωρούμε ότι τίθενται θέματα άρχης. Για ορισμένα τέτοια θέματα μπορεί να μην είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμβασμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Κώστα για αυτήν την εισαγωγή. Ως πρώτος όδης, ε, η κυρία Ιβάνα Μάλετιτς. Όπως πολλά σωστά είπε ο εισηγητής, πρέπει να συμφωνήσουμε σε πολλά πράγματα στην αυριανή μας συνάντηση. Να τονίσω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει η πολιτική συνοχής και οι οικονομικές πολιτικές μονίμως να τις έχουμε στο μυαλό μα παράλληλα. Δεν μπορούμε να τι διαιρέσουμε, γιατί και οι δύο τον ίδιο σκοπό επιδιώκουν ε, βιώσιμα ε, δημόσια οικονομικά, βιώσιμη οικονομική πολιτική και καλή οικονομική και περιφερειακή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε για την διασύνδεσή τους ανάμεσα στην δηλαδή, πολιτική συνοχή και στην οικονομική πολιτική. Και πολλοί από του συναδέλφου με τι τροπολογίε του ακριβώ αυτό θέλουν να επιδιώξουν. Αυτή τη σχέση των δύο πολιτικών. Και ελπίζω στην αυριανή συνάντηση με τον εισηγητή να μπορέσουμε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Η πολιτική συνοχή θα πρέπει να υποστηρίζει την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και των ειδικών αναχώρασης τάσεων και θα πρέπει επίση και το αντίθετο. Ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο θα πρέπει να έχει ως στόχο να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την, ε, το διοικητικό δυναμικό και την εφαρμογή των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων που πάνε χέρι-χέρι με την καλή απορρόφηση και τη σωστή εφαρμογή των, ε, της πολιτικής για τη συνοχή. Πολλές μελέτες ακριβώς αυτό δείχνουν. Όταν ε, διάβασα τις τροπολογίες, ε, βλέπω ότι υπάρχουν πολλές διαφορές ε, μεταξύ των συναδέλφων για τη συγχρηματοδότηση, όπως είπε και ο συγητής. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι μία πηγή χρηματοδότησης μόνο. Έχουμε διάφορες πηγές χρηματοδότησης όμως σε διάφορες χώρες και τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι μία από αυτές τις πηγές και θα πρέπει να είναι τμήμα ενός εθνικού σχεδιασμού ε, με σκοπό την ανάπτυξη. Δεν μπορούμε να διαιρούμε τα επιχειρησιακά προγράμματα ή τη συμφωνία εταιρική σχέσης και τους στόχους που θέτουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, θα πρέπει να ε, διαφοροποιούμε τα προγράμματα εταιρική σχέσης από τις μεταρρυθμίσεις και τα προγράμματα σύγκλησης. Αυτά πρέπει να τα διασυνδέσουμε όλα. Όλες οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όλες τις πηγές χρηματοδότησης, να τις αξιοποιούν και να πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση και να μην χρησιμοποιούμε τα λεφτά του προπολογισμού για τον σκοπό Χ και τα ευρωπαϊκά ταμεία για τον αντίθετο σκοπό. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμπληρωματικότητα. Και ακριβώς γι' αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να αποκλείσουμε την εθνική συγχρηματοδότηση από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Εάν τα ευρωπαϊκά ταμεία είναι τμήμα των εθνικών πολιτικών, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το ξανασυζητήσουμε. Επίσης, ε, σημειώνω ότι κάποιες αντιστροπολογίες υπάρχουν ήδη, έχουν ενσωματωθεί ήδη ε, στην έκθεση του Τόμας Ντόιτς από την ε, Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Περιφερειακή Επιτροπή, εν και ίσως, συνάδελφοι, θα μπορούσατε να δείτε πώς θα μπορούσατε να συνδυαστείτε με την έκθεση ε, Deutsch. Ευχαριστώ. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για κύριος Οζότ. Η συζήτηση για το επενδυτικό σχέδιο δημιούργησε, όπως αναμενόταν, προκάλεσε πολλές τροπολογίες, αναμενόμενο. Καλό θα ήταν να έχουμε μια οριζόντια προσέγγιση στο θέμα των επενδύσεων. Δεν θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε το βασικό στόχο της πολιτικής συνοχής και των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη-μέλη. Η πολιτική συνοχής υποτίθεται ότι μειώνει τις ανισότητες στην ανάπτυξη μεταξύ των διαφορετικών χωρών και των διαφορετικών περιοχών και περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως μπορεί να επηρεάσει την οικονομία Βεβαίως δεν είναι μακροοικονομικό εργαλείο και δεν αντικαθιστά τις ε, εθνικές μεταρρυθμίσεις σε καμία περίπτωση. Εάν οι κυβερνήσεις δεν μπορέσουν σε εθνικό επίπεδο ε, να τα πάνε καλά μακροοικονομικά, οι πολιτικές συνοχής δεν υπάρχουν εκεί για να στηρίξουν ας πούμε, τις κυβερνήσεις εκεί που απέτυχαν. Επομένως θα υποστηρίξω όλες τις τροπολογίες που προωθούν αυτή την άποψη. Τώρα για την παράγραφο 5, εγώ δεν έχω υποβάλει τροπολογία εκεί, αλλά πολλοί άλλοι συνάδελφοι υπέβαλαν. Υποστηρίζω την, τον αποκλεισμό της συγχρηματοδότησης του ΕΦΙΣ από την, τον υπολογισμό του ελλείμματος των κρατών μελών. Επίσης πιστεύω στην ε, εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα και στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν επιλέγουμε έργα, project, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν προωθούμε μια διαδικασία όπου απλώς μετακινούμε χρήματα από τον ένα τομέα στον άλλο. Θα πρέπει να έχουμε ένα πραγματικό ε, σχέδιο συνεργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για αυτά τα δημόσια έργα που χρειάζεται η οικονομία μας. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την τεχνητή διαίρεση των ευρωπαϊκών κρατών σε ή μάλλον των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά ε, κράτη, δηλαδή δεύτερης ε, σημασίας. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη νομοθεσία, αλλά δεν θέλω μεγαλύτερη ολοκλήρωση η εμβάθυνση της Τραπεζικής Ένωσης. Παρά τα όσα είπε ο εισηγητής, νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για να προκύψει ένα καλό κείμενο μέσα από όλα αυτά, μέσα από όλες αυτές τις διαφορές. Ευχαριστώ Στανισλάβ. Δεν βλέπω κανένα από την Άλντε, ούτε την Παλώμα από την Κούε, ούτε άλλο πρόσωπο της ε, Κούε. Οπότε, ο Ένεστ, Ουρτασούν, των Πρασίνων. Όπως είπα και την προηγούμενη φορά, το κείμενο μας ε, φαίνεται καλό. Νομίζω ότι συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα έπρεπε να είναι. Θα αναφερθώ σε ορισμένες τροπολογίες που υποβάλαμε και που θεωρώ σημαντικές και όπως είπε και ο εισηγητής προηγουμένως θα πω ότι για ποια σημεία υπάρχουν δυσχέρειες για την ομάδα μου για να έχει στοιχείο ο για την αυριανή συνεδρίαση. Νομίζω πως θα ήταν σκόπιμο όταν μιλάμε για το σχέδιο Juncker να έχουμε πιο ουδέτερη διατύπωση, τροπολογία 31. Νομίζω ότι είναι καλό να έχουμε ουδέτερη διατύπωση, όπως επιτύχαμε σε άλλα σημεία. Σε ορισμένα άλλα σημεία θέλουμε να καθορίσουμε καλύτερα πώς θα πρέπει να γίνεται η επιλογή των προγραμμάτων του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει δηλαδή ορισμένα να εξαιρούνται μέσω crowding out και θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτά τα οποία έχουν ε, κοινωνική και περιβαλλοντική θετική επίπτωση. Αναφέρομαι επίσης στην τροπολογία μας 64 όπου τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ κρατικών φορέων και του ΕΦΣΥ είναι σημαντικό αυτό ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο οι εθνικοί φορείς και όπω είπαν και άλλοι νομίζω ότι η εξαίρεση της χρηματοδότηση από την εφαρμογή του ελλείμματος, από τον υπολογισμό του ελλείμματο είναι σημαντική. Αυτό που λέει το 56. Από τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Ορισμένοι λένε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το κοκτέιλ ε, δημοσιονομική εξυγίανση και διαστροτικές μεταρρυθμίσεις για ορισμένε περιφερειακές χώρες πολλές από τις προσπάθειες που κάναμε μέσω της πολιτικής συνοχής καταστράφηκαν λόγω των αυτοκτονικών πολιτικών ε, δημοσιονομικής εξυγίανσης θα ήταν λάθος λοιπόν να συνεχιστούν τέτοιες πολιτικές. Ενώ ακριβώς θέλουμε η έκθεση να τονίσει πώς θα προωθήσουμε την κοινωνική και εδαφική συνοχή. Νομίζω ότι οι τροπολογίες αυτές πρέπει να συμπεριληφθούν. Και υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες άλλων ομάδων που είναι πολύ θετικέ κατά τη γνώμη μα και μπορούμε να στηρίξουμε. ορισμένε που τονίζουν ότι κάποια προγράμματα μπορεί να είναι συμπληρωματική επιβάρηση του προπολογισμού. Υπάρχει μια καλή τροπολογία των φιλελεύθερων επ' αυτό. Είναι μια πρόταση του Χώνας Φερνάντε, των σοσιαλιστών που λέει να δούμε αν μπορεί να υπάρχει ένα σύστημα επιδομάτων ανεργίας που να βασίζεται σε αυτό. Αυτά είναι γενικά αυτά που θέλουμε να προτείνουμε στη συνεδρίαση αύριο των συντονιστών και που θα ήθελα να τα ξέρει ήδη ο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είδα ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν σημειώνει με ζήλο τα όσα ακούει. Επιθυμείτε να τοποθετηθείτε. Ορίστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. συμφωνούμε με τις περισσότερες από τις τοποθετήσεις που ακούσαμε. Κάποιες ενστάσεις έχουμε απέναντι στο επιχείρημα ότι εάν οι κυβερνήσεις δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους στις ε, πολιτικές συνοχής. Νομίζουμε ότι στις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους η πολιτική συνοχής στήριξε χώρες με δημόσιο χρέος μειώνοντας ε, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και αν δείτε και την έκθεση, την πρώτη σελίδα της έκθεσης συνοχής θα δείτε ότι αναφέρεται στην επίπτωση της πολιτικής συνοχής στις χώρες μέλη. Και ίσως κάτι ακόμη. Αυτό, αυτό όμως είναι το βασικό επιχείρημα. Βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις ό,τι αφορά την έκθεση συνοχής, πολύ ευχαρίστως να απαντήσω. ο Προεδρεύων κ. Σίμων. Ας λάβει το λόγο πάλι λοιπόν ο εισηγητής ε, κ. Μαυρίδης. Ευχαριστώ. Σύντομο σχόλιο. Όλοι συμφωνούμε νομίζω πάνω σε μια πτυχή της γνωμοδότησης ότι οι πολιτική συνοχής και οι οικονομικές πολιτικές βεβαίως βαίνουν παραλλήλως. Νομίζω όμως ότι εκεί όπου αρχίζουν να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις είναι σχετικά με το σε ποιο βαθμό η πολιτική συνοχής θα πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς σαφή σύνδεσμο με εξειδικευμένες προϋποθέσεις σχετικά με την εθνική οικονομία. Αν όλοι συμφωνούμε ότι η αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι το ουσιώδες περιεχόμενο της πολιτικής συνοχής. Αυτό είναι βέβαια ένα πράγμα το οποίο μας αποτρέπει από το να επιβάλλουμε κάποιες συγκεκριμένες μακροοικονομικές προϋποθέσεις. Άκουσα βεβαίω όλες τις απόψεις και είμαι βέβαιος ότι αύριο θα διεξαχθεί επικοδομητικός διάλογος και θα συνεχίσουμε μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιγητά. Στις 20 Απριλίου θα ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή Οικονομικών η ΔΕ Επιτροπή Ρέγγι 4 5 Μαΐου. Εδώ λοιπόν κλείνει η συζήτηση αυτού του θέματος. Πηγαίνουμε στο υπαριθμό 10 διάφορα, δεν υπάρχουν εδώ διάφορα. Και το 11 διακόπτω την συνεδρίαση. Το 11 είναι μονάχα ότι θα ξαναειδωθούμε στις 20 Απριλίου μεταξύ και 18 και 30 ώρων. Ευχαριστώ και είστε